Ε, Ο πρόεδρος Ρεμπέλο Ντε Σόζα, πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την ε, υποδοχή που μας επιφυλάξατε στον πρόεδρο Ρεμπέλο Δε Σόσα της Πορτογαλίας. Θα ήθελα να σας πω κύριε πρόεδρε, όχι μονάχα καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά καλώς ήλθατε με μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί κυρίες και κύριοι, μετά από την τις εκλογές και την ανάληψη της εξουσίας από τον κύριο Ρεμπέλο Δεσόσα πήρα τηλέφωνο για να τον συγχαρώ και του είπα το εξής. Θα ήθελα, μου είπατε, τότε η πρώτη μου επίσκεψη στην, ε, ως πρόεδρο της Πορτογαλίας να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι μονάχα μια συμβολική χειρονομία του Προέδρου της Πορτογαλίας, αλλά είχαμε και μια πολύ έντονη συζήτηση και ενδελεχή για τον ρόλο της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν μπορώ να σας παραθέσω, είπατε ότι η επίσκεψή σας εδώ είναι και έκφραση της βαθιάς ευρωπαϊκής μου πεποίθησης και θέλω να το γνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Πορτογαλία έχει ένα πρόεδρο ο οποίος θέλει να εργαστεί εντατικά για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και θέλει να συμμετάσχει απόλυτα στο ρόλο της Ευρώπης στην διεθνή σκηνή. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας και σας δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την τιμή που μου κάνετε να με προσκαλέσετε στο σπίτι της Δημοκρατίας ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε Μάρτιν Σούλτς, για το γεγονός ότι έχω την ευκαιρία να λάβω το λόγο ενώπιον των εκλεγμένων εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Λαού και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι το σπίτι της δημοκρατίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κλίμακα που εδράζεται στις αρχές της ελευθερίας, της ασφάλειας, του ουμανισμού, της συμμετοχής των πολιτών από την συνέλευση αυτή και ο κάθε ένας από εσά είναι ένας εγγυητής αυτών των αρχών. Το να μπορώ να είμαι εδώ σήμερα είναι και μήνυμα και ένα μήνυμα για τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για την ε, επαν, επανέλευση και την εδραίωση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Είναι και σήμα μιας προσωπικής δέσμευσης που ξεκίνησε από μια πολύ παλιά πορεία της χώρας μου. Ανήκω σε μια γενιά Πορτογάλων για τους οποίους η, η στην Ευρώπη ήταν ένα όραμα το οποίο ήταν αδιάσπαστο από την έννοια της δημοκρατίας, της αποαπικιοποίησης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η μεταβολή από, δημο, δικτατορία σε δημοκρατία στην Πορτογαλία πέρασε από το τέλος της αυτοκρατορίας μας αλλά όχι και από το τέλος της θέλης Πορτογαλίας να παραμείνει μέσα στην Ευρώπη που είναι το γεωγραφικό της λίκνο. Μετά από την δεκαετία των 60 του προηγούμενου αιώνα η Ευρώπη ήταν και ο χώρος προς τον οποίο είχαν κατευθυνθεί περισσότεροι μετανάστες από την Πορτογαλία καθώς και το εμπόριο της Πορτογαλίας. Εμείς πιστεύουμε στην Ευρώπη γιατί είναι παράδειγμα ειρήνης, αλληλεγγύης, ανάπτυξης, κοινωνική ισότητα πολιτισμικού χώρου αλλά επίσης για μας υπήρξε και το κίνητρο και το έναυσμα για τη δημιουργία μιας νέας Πορτογαλίας. Γι' αυτό θέλω να υπενθυμίσω με μεγάλη νοσταλγία το πρώτο μου ταξίδι μαζί με μια αντιπροσωπεία πανεπιστημιακών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πιο δύσκολη περίοδο της Πορτογαλικής Επανάστασης. Ή επίσης θέλω να υπενθυμίσω και την επιρροή της Ευρώπης στην δραστηριότητά μου 20 και περαιτέρω χρόνια ως βουλευτή στην ξεκινώντας με την πρώτη συντακτική συνέλευση Πορτογαλίας το 1975-1976. Γι' αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική η αίτηση ένταξη τη Πορτογαλίας το 1977 που οδήγησε σε μακρέ διαπραγματεύσει μέχρι το 1985 και επίσης η διαδικασία, η δύσκολη διαδικασία που οδήγησε στο ενιαίο νόμισμα όταν εγώ ως ηγέτης της αντιπολίτευσης υποστήριξα τρεις κρατικούς προϋπολογισμούς για μέσα σε μια μειονοτική κυβέρνηση και έτσι μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε την είσοδο της Πορτογαλίας στη ζώνη του ευρώ. Θα ήθελα επίσης να σας ε, ομολογήσω την χαρά και την ε, ε, υπερηφάνεια που ένιωσα όταν ένας Πορτογάλος, ο Ζωζέ Μανουέλ Ντουράου Μπαρόσο, έγινε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης νιώθω ιδιαίτερη η περηφάνεια για το έργο των Πορτογάλων βουλευτών από όλες τις παρατάξεις σε αυτήν την ίδια συνέλευση που βρίσκομαι σήμερα. Οι πεπιθήσεις μας από το παρελθόν είναι στεναρέ και δεν αλλάζουν. Συνεχίζω να είμαι πεπισμένο για την απαράγραπτη σημασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ευρώπη και τον κόσμο. Εμεί από τότε που είμαστε δημοκρατικό χάρτο ω Πορτογαλία συνεχίζουμε να ακολουθούμε την εθνική στρατηγική. Όλοι οι πρόεδροι και όλε οι κυβερνήσει έχουν ακολουθήσει αυτή την πορεία. Η Πορτογαλία βρίσκεται σήμερα εφέτος στα 40 χρόνια του συντάγματός της και του συντάγματο αυτού που ήταν ο οδηγό χάρτη για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Πορτογαλία. Την εδραίωση αυτή τη δημοκρατία στην Πορτογαλία η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, οι ευρωπαϊκέ κοινότητε έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο. Ήταν πάρα πολύ σημαντική και εξακολουθεί να είναι η συνεισφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη τη χώρα μου, για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των πολιτών μα η Πορτογαλία μπόρεσε με μεγάλη επιτυχία να χρησιμοποιήσει τα διαφθορτικά κονδύλια τα οποία ήρθαν από την Ευρώπη. Εξυγχρόνισε τον παραγωγικό τη ιστό. Έκανε καλύτερα εκπαιδευμένα το εργατικό της δυναμικό. Βελτίωσε τι βασικές υποδομέ. Αλλά για να μπορέσει να προσαρμοστεί στου ευρωπαϊκού κανόνε, η Πορτογαλία χρειάστηκε να κάνει σε 12 χρόνια αυτό που οι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, οι πιο ισχυρέ οικονομίε, είχαν κάνει σε πάνω από 40 χρόνια. Και κατάφερε λοιπόν να επιτύχει την αποαπικιοποίηση σε δύο χρόνια, να υποδεχθεί 700.000 9.700.000 ε, Πορτογάλους και επίσης Αφρικανούς που ήταν Πορτογαλόφωνοι στο εδαφός της είδε να συνεχίζεται έμεσα η στρατιωτική εξουσία μέχρι το 1982 κατάφερε να ξεφύγει από μια εν μέρη αγροτική, απικιακή και κλειστή οικονομία προς μια ευρωπαϊκή παγκοσμιοποιημένη οικονομία και ανοιχτή. Σιγά σιγά πέρασε στην ε, επανιδιωτικοποίηση αυτής της ε, οικονομίας με βάρος ειδικό στις υπηρεσίες και τις νέες βιομηχανίες. Το τίμημα αυτών των αλλαγών σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ήταν πολύ σημαντικό. Χωρίς την χρήση των κοινωνικών ταμείων που έδειξαν την κατανόηση και την υποστήριξη της Ευρώπης προς την Πορτογαλία θα ήταν αδύνατο να επιτύχουμε την απαραίτητη αυτή εδραίωση και παγίωση με τις ε, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κρίσεις του 2008 και του 2009 προσθέθηκαν προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα διαρθωτικά προβλήματα στην Πορτογαλία και για 3,5 χρόνια έλαβε χώρα ένα πρόγραμμα προσαρμογής όπου έλαβε μέρος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ενέργειες αυτές έθεσαν σε δοκιμασία την ιστορική ικανότητα των Πορτογάλων να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις και να προβαίνουν σε προσωπικές θυσίες ώστε να μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι δημοσιονομικές ισορροπίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας μας. Ως πρόεδρος τη Πορτογαλικής δημοκρατία νιώθω μεγάλη η περηφάνεια που μπορώ να είμαι σήμερα ενώπιον της ε, συνέλευσής σας και, να μπορέσω, και του, του γεγονότος ότι μπορώ να σας πω ότι η Ευρώπη δεν παρέλειψε να βοηθήσει την Πορτογαλία. Και η Πορτογαλία τίμησε απόλυτα τις δεσμεύσεις της και μπόρεσε να εξέλθει με καθαρό τρόπο από το πρόγραμμα ε, σταθεροποίησης και προσαρμογής. Σήμερα η Πορτογαλία εξακολουθεί και θέλει να εξακολουθήσει να εγγυάται για τις δημοσιονομικές ισορροπίες, για τον έλεγχο του ελλείμματός τους, για το έλεγχο του δημόσιου χρέους της και συγχρόνως θέλει να ξεκινήσει να δίνει πάλι βοήθεια στους κοινωνικούς τομείς οι οποίοι ήταν τα πιο μεγάλα θύματα του άμεσου παρελθόντος. Πιστεύουμε ότι πέραν από τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις εξαγωγές είναι απαραίτητο να ευνοήσουμε την κατανάλωση των οικοκυριών για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη είναι ένας δρόμος που στοχεύει στους ίδιους μακροοικονομικούς και δημοσιονομικούς στόχους, αλλά που εν μέρει είναι διαφορετικός από τον ε, παλαιό. Ε, καθοδηγείται από μια κυβέρνηση ευρωπαϊκή που σέβεται τους διεθνούς, ε, τις διεθνείς δεσμεύσεις που υποστηρίζεται στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο από μία από τις δύο κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες, αλλά και από κόμματα άλλη σημαντική ευρωπαϊκή οικογένεια που μέχρι τώρα ήταν εκτός του τομέα της ε, συνταγματικής εξουσίας ε, της, ε, της Πορτογαλίας ακόμα και με ρίζες που έρχονται από διαφορετικά δόγματα από αυτά στα οποία εντάσσεται η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως πρόεδρος όλων των Πορτογάλων αισθάνομαι πως είναι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή να, να, να ηρεμήσουμε, να αποδραματικοποιήσουμε να επουλώσουμε πληγές και να οικοδομήσουμε συνενέσεις. Το μήνυμά μου είναι λοιπόν σαφές, ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, σταθερότητα, άρνηση των πολιτικών κρίσεων, ε, ξεκινώντας από τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα, αναζήτηση διευρυμένων συγκλήσεων, η ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και μάλιστα έγινε πρόσφατα ένα θετικό βήμα ε, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε βελτίωση των τοπικών αρχών, των ε, διοικητικών αρχών, ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη. Και πραγματικά εύχομαι ε, ειλικρινά να έχουμε πλήρη επιτυχία στην απαιτητικό δρόμο της δημοσιονομικής ρύθμισης, της λιτότητας, αλλά και των κοινωνικών ανησυχιών που έλειπαν ε, περισσότερο από τον δυναμισμό αυτής της εσωτερικής αγοράς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαι ένας αδιόρθωτος ευρωπαϊστής. Η Ευρώπη ε, που ονειρευόμουν και ονειρεύομαι και την οποία ονειρεύεται και η μεγάλη πλειοψηφία των Πορτογάλων αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις πολύ πιο περίπλοκες από αυτές που ε, αντιμετώπισε στο παρελθόν. Αυτές οι προκλήσεις μας λένε πως δεν είναι τώρα ο καιρό να αμφισβητήσουμε ή να ε, διστάσουμε. Ε, ο προβληματισμός σε σχέση με το μέλλον της Ένωσης θα πρέπει να δώσει μια νέα ζωή σε ένα μοντέλο της Ευρώπης που ζει σε μια περίοδο ειρηνική ε, και ευημερή. Ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε απομακρύνοντας ε, ξενοφοβικές ε, συμπεριφορές, καταπολεμώντας υπερβολικούς εθνικισμούς, απορρίπτοντας τους στήρους σοβινισμούς, αρνούμενοι από μονατισμούς ξεπερασμένους. έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα τεράστιο και αξιοζήλευτο μέλλον, και, αλλά και κληροδότημα ε, η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι καρποφόρα μόνο εφόσον υπάρχει μόνιμος και διαρκής διάλογος με τους Ευρωπαίους πολίτες, ε, σεβόμενοι τις θεμητές τους προσδοκίες να ζουν σε ένα χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, ανάπτυξης, απασχόλησης, ευημερίας και αλληλεγγύης. Και γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό οι Ευρωπαίοι και οι εθνικοί ηγέτες να προσέχουν σε αυτές τις προσδοκίες, να προσέχουν και να ε, ακούν, να φουγκράζονται την δηλωμένη βούληση των δημοκρατικών μας κοινωνιών. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παιδαγωγική ε, και στην προσέγγιση εγκύτητα με τους πολίτες. Η Ευρώπη που εγώ ονειρεύομαι μένει ενωμένη και αλληλέγγυη. Ε, προσέχει τις πιθανές ε, αφήξεις ε, καλύπτοντας τις πιθανές αφήξεις ε, αλλά χωρίς αναχωρήσεις, ε, αναζητώντας πάντοτε κοινέ λύσεις για να καλυφθούν ο αντίκτυπος και οι επιπτώσεις των κοντινών πολέμων. Το θέμα το προσφυγικό, η Πορτογαλία δώσε το παράδειγμα σε αντιστοιχεία, σε αναλογία με τον πληθυπισμό μας, έχουμε αποτελέσει τον μια κύρια χώρα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που δείξαμε διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε πρόσφυγες στο πλαίσιο της ε, πορτογαλικής κοινότητας. Situação esta que είναι τέτοια η κατάσταση που απαιτεί οι ουσιαστικές, τα ουσιαστικά ζητήματα να μην ξεχαστούν με, μέσω βραχυπρόθεσμων απλών συμφωνιών που όλοι επιθυμούμε ότι δεν θα αποδεχθούν αμφισβητήσιμες ή ανεπαρκείς. Η Ευρώπη που εγώ ονειρεύομαι, που ε, θριάμβευσε πολλές φορές απέναντι στους βαρβάρους και στους απολυταρχισμούς, ήταν πάντοτε αυτή που μπορεί να νικήσει τις ε, απειλές του θρησκευτικού φανατισμού, του πολιτικού φανατισμού και της τρομοκρατίας. Γι' αυτό μόνο και ε, δρώντας αλληλέγγυα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές και εδώ ακριβώς εκφράζω εκ νέου την αλληλεγγύη μου με τη Γαλλία και με το Βέλγιο. Η Ευρώπη που εγώ ονειρεύομαι φιλοδοξεί να έχει πραγματικό παγκόσμιο πολιτικό αντίκτυπο. Αντίκτυπο που θα είναι ανάλογος με το εμπορικό της βάρος. Είναι σημαντικό να μπορούμε να ηγούμαστε σε, παγκόσμια ζητήματα όπως ε, τη διαφάνεια στη ε, χρηματοπιστωτικά ε, θέματα ώστε να υπάρχει διαφάνεια καθώς και στην δικαιοσύνη την περιβαλλοντική. Εγώ ονειρεύομαι μια Ευρώπη που θα θελήσει να ακολουθήσει την πολιτική και το δικαίωμα, αλλά ταυτόχρονα θα συμβαδίζει με το ρυθμό της επιστημονικής, τεχνικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής πραγματικότητας. Μια Ευρώπη που θα μπορέσει να καλύψει τα όνειρα των ε, ψηφοφόρων, των νέων, των ξεχασμένων που αγωνίζονται με ενάντια στην απεσιοδοξία. Η Ευρώπη που εγώ ονειρεύομαι έχει στην Πορτογαλία μία τεράστια, μία μεγάλη απεριόριστη λεγεώνα ε, ε, ανθρώπων που ονειρεύονται για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την ελληνική, τη διαφάνεια και την ε, λαϊκή στήριξη. Η Ευρώπη που ονειρεύομαι έχει στην Πορτογαλία στο μέτωπο αυτού του αγώνα ε, πολλούς αισιόδοξου ανθρώπους. Ε, διαφορετικά δεν θα είναι πια το μέλλον η Ευρώπη. Η Ευρώπη που εγώ ονειρεύομαι διατηρεί στη μνήμη της αυτό που η Πορτογαλία με τη δύναμη της απλότητάς της έφερε από άλλες ε, υπήρους πολιτισμούς και πολιτισμούς ε, και αυτό μας πλουτίζει τόσο πολύ. Η Πορτογαλία που φέρνω μαζί μου σήμερα έχει διασχίσει θάλασσες και ωκεανούς, αλλά ποτέ δεν ξέχασε ότι ανήκει στην γη του Όμηρου, του Σέξπιρ, του Γκέτε, του Προύς, του Θερβάντες, του Δάντη, του Τζόις, του Στρίντμπεργκ, του Κούντερα, του Κάφκα, του Ζιμπόρσκα και αλλά και του Πεσόα τη Ζιμπόρσκα, αλλά και του Πεσόα. Εμείς είμαστε όλοι Ευρωπαίοι και πάντοτε θα είμαστε Ευρωπαίοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Ε, ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Καλή επιτυχία. Σας ευχόμαστε στην ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, είστε πρόσδεκτος πάντοτε και πραγματικά η ομιλία σας ενθάρρυνε όλους όσους αυτό το σώμα σκέπτονται όπως εσείς και όπως είδατε είναι η συντριπτική πλειοψηφία. chiedere la parola. Buongiorno, colleghe e colleghi. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε τις ε, ψηφοφορίες, αλλά ζητά τον λόγο ο κύριος Βάγκελ. Παρακαλώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Το κοινοβούλιο αυτό το, ψήφισε ένα ψήφισμα σε σχέση με την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Στο κεφάλαιο 78 αυτού του ψηφίσματος έχουμε το θέμα των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Γίνουμε το αίτημα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σαχέλ. Ε, υπήρξε μια απεργία πείνας νέων στο Μαρόκο που καταδικάστηκε αδικαιολόγητα από δικαστήριο του Μαρόκο. Θα ήθελα να απευθυνθώ εδώ στο σώμα ούτω ώστε να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές στο Μαρόκο και να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωση των κρατούμενων και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στις ψηφοφορίες.